Κυρίε και κύριοι, Στι 24 Ιουλίου έγινε ένα φρικτό ατύχημα στο Σαντιάγκο Τε Κομποστέλε. Μετά από αυτό ε, το φοβερό ατύχημα απεβίωσαν 79 άτομα. Και λίγες μέρες αργότερα και στην Ιταλία χάθηκαν ε, 39 άτομα στην καμπανία 39 άτομα χάθηκαν σε ένα ατύχημα λεωφορείου μας σόκαραν όλα αυτά τα ατυχήματα και θα ήθελα εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκφράσουμε τη θλίψη μας και τη συμπαθιά μας και τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες όλων των θυμάτων Τώρα μέχρι τις ευρωπαϊκές εκλογές μας έχουν μείνει οκτώ μήνες. Οκτώ μήνες κατά τους οποίους εμείς θέλουμε να κινητοποιήσουμε τους ευρωπαίους πολίτες να έρθουν στις ευρωπαϊκές εκλογές, να συμμετάσχουν σε αυτές τις εκλογές ενεργά. Για αυτούς τους 8 μήνες, αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε αρκετά έργα τα οποία πρέπει να ολοκληρώσουμε και ξέρουμε ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει πολλά τα τελευταία χρόνια. Η δική μας θητεία είναι ιδιαίτερα φιλόπονη θητεία και είχαμε πολύ καλά επιτεύγματα μέχρι τώρα. Πίσω μας έχουμε πέντε χρόνια κρίσης ε, και δεν μιλά πια κανείς για την υπαρξιακή κρίση του ευρώ το ευρώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση παρόλα αυτά χρειάζονται σταθεροποίηση. Ένα ε, στοιχείο σταθεροποίησης ε, είναι η ένταξη της Λετωνίας στη ζώνη του ευρώ την 1η Ιανουαρίου της επόμενης χρονιάς. Η ενεργεία των νέων είναι ένα από τα σημεία που μας απασχολούν και στο πλαίσιο ε, των τωρινών διαπραγματεύσεων των ε, χρηματοδοτικών προοπτικών ε, θα λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα σημεία ώστε να καταπολεμήσουμε την αργία ε, των νέων και να λάβουμε εκ των προτέρων μέτρα υπό τη μορφή του front loading για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ενεργεία των νέων. Αυτό είναι κάτι το οποίο οι αρμόδιες επιτροπές το συζητούν και ελπίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το ίδιο ισχύει και για την Τραπεζική Ένωση. Η Τραπεζική Ένωση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και πιστεύω ότι εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να την υλοποιήσουμε. Και θα φροντίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο για την περαιτέρω εδραίωση τη ε, σταθερότητα στην Ευρώπη. Ε, ελπίζω ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στους επόμενους ε, μήνες θα ολοκληρωθούν όλα τα, όλες τις νομικές πράξεις που απαιτούνται για αυτή την κατεύθυνση. Η ταχεία ολοκλήρωση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου σαφώς είναι ένα κεντρική σημασία ε, πρόγραμμα. Πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές ε, καταλήξαμε σε μια συμφωνία για τα ανώτατα όρια για την επόμενη περίοδο χρηματοδότησης. Και δεν ήταν καθόλου απλό το να καταλήξουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η πλειοψηφία ε, έκανε σημαντικές υποχωρήσεις για να μπορέσουμε να το επιτύχουμε αυτό. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη νομική βάση για το πολιτικό οικονομικό πρόγραμμα και θα πρέπει να συνεχίσουμε για να μπορέσουμε ε, να ψηφίσουμε τον κανονισμό και το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο όταν έχουν τηρηθεί όλες οι προθεσμίες. Ε, προς το παρόν ε, δεν βλέπω να έχουν τηρηθεί όλες οι προθεσμίες. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, το έργο μας και να βρούμε τις κατάλληλες συμβιβαστικές λύσεις. Και τώρα περνώ στην ημερήσια διάταξη για τη σημερινή μας συνεδρίαση. Και χαίρομαι διότι όλοι οι συνάδελφοι είναι σήμερα παρόντες, πολλοί συνάδελφοι που δεν έχω δει πολύ καιρό τώρα και χαίρομαι που συμμετέχουμε όλοι στην επανάληψη της Συνόδου Λομέλειας ε, και χαίρομαι που βλέπουμε και τον πρόεδρο Άλβαρο και πάλι κοντά μας. και θα ήθελα να εκφράσω την ελπίδα ότι ο πιτός συνάδελφός μας Παπαστάμκος ε, ο οποίος πηγαίνει καλύτερα αλλά ακόμη δεν είναι εντελώς καλά, ελπίζω ότι και εκείνο σύντομα θα είναι κοντά μας στη συνεδρίαση και θα μπορέσει και αυτός να συμμετάσχει στη συνεδρίασή μας. Και εκφράζουμε όλες τις ευχές μας προς την οικογένειά του. Καλή ανάρρωση. Τα πρακτικά τη συνεδρίασης του Ιουλίου ε, είναι διαθέσιμα και θέλω να σα ρωτήσω αν υπάρχουν αντιρρήσει ή παρατηρήσει για τα πρακτικά.